okay, you can start. Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Από ό,τι φαίνεται τα τεχνικά θέματα ξεπεράστηκαν. Ελπίζω να μην ξαναπροκύψει κάτι πριν το τέλος της συνεδρίασης. Είναι η τελευταία μας συνεδρίαση πριν τις χριστουγεννιάτικες διακοπές. και θα ξεκινήσω με το πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έγκρισή της. Θα ήθελα στις ανακοινώσεις του Προέδρου να αναφερθώ λίγο στο ΚΑΠΣΑΤ, να σας ενημερώσω για τα τελευταία γεγονότα και βεβαίως να μιλήσουμε λίγο για τη συνέχεια που θέλουμε να δώσουμε και τις πρωτοβουλίες μας σαν Επιτροπή Πολιτισμού. Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο στην ημερήσια διάταξη. Όχι. Ας θεωρήσουμε λοιπόν ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ανακοινώσεις του Προέδρου, σημείο 2 της ημερήσιας διάταξης. Από ποιες γλώσσες έχουμε διερμηνία. Ξέρετε ότι αναμεταδίδεται στο διαδίκτυο η σημερινή συνεδρίαση. Έχουμε επίσης ε, τα πρακτικά της 22ης Νοεμβρίου που εστάλησαν σε όλους τις 24 ε, Νοεμβρίου με mail και θα θεωρήσουμε ότι είναι εγκεκριμένα αν μέχρι τις 28 του μηνός κανείς δεν έχει υποβάλει καμία παρατήρηση ή πρόταση για αλλαγή. Κάψατ ο κανονισμός, κάψατ και θα ήθελα να σας πω κάποια από τα θέματα τα ξέρετε, ξέρετε ότι η Επιτροπή Γιούρη έχει γνωμοδοτήσει για το θέμα αυτό. Πρόκειται για τις ε, εκπομπές ε, τηλεόρασης, ραδιοφώνου και μέσω διαδικτύου. Εγκρίθηκε η Επιτροπή, από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων και όπως ξέρετε σύμφωνα με τον κανονισμό, σύμφωνα με το άρθρο 54, σύμφωνα με το άρθρο 69C υπάρχει κατανομή αρμοδιοτήτων και βεβαίως έχουν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ όλων των πολιτικών ομάδων και μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στη Μήνη Ολομέλεια αποφασίστηκε να υπάρξει αυτή η διαπραγμάτευση και μέχρι τις 12 Δεκεμβρίου στην επόμενη Ολομέλεια να ολοκληρωθεί ο κύκλος των διαπραγματεύσεων. Οι ειρηνικέ αυτές ε, διαπραγματεύσεις όμως δεν προχώρησαν, γι' αυτό και μιλάμε σήμερα για μια νομική πράξη και τον Ιανουάριο στην Ολομέλεια σε μια πρώτη ανάγνωση θα συζητηθεί το θέμα αυτό. Οι τροπολογίες μέχρι τις 10 Ιανουαρίου του 2018 στις 12 το μεσημέρι μπορούν να υποβληθούν. Εμείς λοιπόν θα συνεδριάσουμε 22 και 23 Ιανουαρίου για πρώτη φορά τον επόμενο χρόνο. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω ότι ουσιαστικά σήμερα θα πρέπει να δούμε λίγο σύμφωνα με το άρθρο 54 του κανονισμού αν πρέπει εμείς να υπερασπιστούμε αυτό το άρθρο 54 και βεβαίως οι διάφορες διαπιστώσεις ε, της έκθεσης της Επιτροπής ε, Νομικών Υποθέσεων δεν ε, συμβαδίζει με την δική μας νομοδότηση, αυτή δηλαδή που με μεγάλη πλειοψηφία ψηφίσαμε εδώ. Έχουμε λοιπόν τρεις δυνατότητες και θα ήθελα να σας τις παρουσιάσω. Καταρχήν, θα μπορούσαμε σήμερα να κάνουμε μια πρώτη απόφαση που στην περίπτωση αυτή υπάρξει, στην περίπτωση συγγνώμη, που υπάρξει απόρριψη της σημερινής πρότασης από την Ολομέλεια. Και υπάρχουν εδώ οι συγκεκριμένες προτάσεις, η 1.19, 21, 119, οι οποίες αποφασίστηκαν στη δική μας γνωμοδότηση τον Ιούνιο και να θέσουμε αυτά τα σημεία στην Ολομέλεια σε ψηφοφορία. Νομίζω ότι η Γραμματεία έχει εντοπίσει όλα αυτά τα σημεία λέγοντας ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη στην έκθεση της νομικής επιτροπής. Και βεβαίως επειδή υπάρχει κατανομή των αρμοδιοτήτων, έχουμε δικαίωμα να υποβάλουμε αυτά τα σημεία. Βάσει της ε, κατανομής των αρμοδιοτήτων μπορούμε να μην, ε, και αυτή είναι η δεύτερη εναλλακτική, να μην πάρουμε τέτοια προαπόφαση σήμερα, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε να υπάρξει μια δική μας συνεδρίαση της Επιτροπής μας, δηλαδή πριν την 10η Ιανουαρίου και να συζητήσουμε το άρθρο αυτό 54, τρίτη εναλλακτική να δεχτούμε την πρόταση της Επιτροπής Γιούρη και να μην επανέλθουμε στο θέμα των αρμοδιοτήτων τις οποίες μοιραζόμαστε με τον Πηγιούρη. Εγώ πραγματικά θεωρώ ότι από τη στιγμή που έχουμε πολύ σημαντικά αν θέλετε σημεία στα οποία θέλουμε να λάβουμε υπόψη στην τελική έκθεση, χωρίς βεβαίως να ζητήσουμε εδώ αντιπαράθεση. Και εγώ σαν εισηγήτρια, αλλά και άλλα μέλη της Επιτροπής, νομίζω θεωρούν ότι με πολύ δημοκρατικό τρόπο επεξεργαστήκαμε όλα αυτά τα θέματα, ότι Πρόκειται για μια νομοθετική διαδικασία και σαν Επιτροπή Πολιτισμού έχουμε συγκεκριμένες αρμοδιότητες και δικαιώματα. Αυτό που ζητάμε δηλαδή είναι απρός να υπερασπιστούμε την απόφαση που πήραμε μετά από συζήτηση και αυτή τη δημοκρατική διαδικασία. Από τη στιγμή λοιπόν που θα προχωρήσουμε με αυτήν τη συγκεκριμένη θέση, οι διαπραγματεύσεις θα ξεκινήσουν, όπως είπαμε μετά τις 10 του μηνός και το ερώτημα είναι τι θέλετε να κάνουμε για μένα τουλάχιστον. Πρέπει να εγγυηθούμε και να προσπιστούμε τα δικαιώματα της Επιτροπής Πολιτισμού. Έχουμε ε, και εμείς αρμοδιότητες ε, μαζί με την Επιτροπή Γιούρη Σύμφωνα λοιπόν και με την ανάλυση της γραμματείας, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εδώ να απορρίψουμε αυτή την εντολή. Υπάρχουν οι συγκεκριμένες τροπολογίες, όλα αυτά τα σημεία τα οποία σας τα προανέφερα, μπορούμε να τα επανυποβάλουμε στην Ολομέλεια έτσι ώστε να εγγυηθούμε και να ε, υπερασπιστούμε τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Πολιτισμού. Εγώ δηλαδή προσωπικά είμαι υπέρ της εναλλακτική 2. Βεβαίως δεν ε, υπάρχει λιμένη απόφαση. Στις 10 ε, του μηνός ε, θα μπορούσαμε να συναντηθούμε. Εγώ θα ήθελα με τα μέλη της ε, πολιτικής μου ομάδας να συζητήσουμε το θέμα, να αποφασίσουμε, να ψηφίσουμε. Και δεν είναι μόνο οι τροπολογίες της Επιτροπής Πολιτισμού. Υπάρχουν και κάποιες άλλες τροπολογίες που μπορεί να υποβάλουν οι πολιτικές ομάδες που έχουν υποβάλει, που θέλουν να τις ε, υπερασπιστούν. Νομίζω λοιπόν ότι αφού δεν μπορέσαμε με άλλο τρόπο να προχωρήσουμε, ναι, εναλλακτική 2 και ίσως ε, να συζητήσουμε το θέμα την Ολομέλεια, πριν την Ολομέλεια η Δευτέρα ή την Τρίτη. Πρόεδρος. Το θέμα είναι ότι η πρώτη εβδομάδα που θα επανέλθουμε το 2018 να δουλέψουμε είναι ομάδα ε, πολιτικών ομάδων και μόνο τη Δευτέρα ενδεχομένως θα έχουμε χρόνο. Ναι, Ξέρετε τα πράγματα όμως πώς είναι. Μετά τις διακοπές δεν εμφανίζεται κανείς εδώ τη Δευτέρα. Τι να πω. Ναι, εντάξει, εγώ άμα θέλετε να ξεκινήσουμε με την χρονιά μας, τη σεζόν μας, της Επιτροπής Πολιτισμού με ενθουσιασμό. Την Τρίτη δεν θα έχουμε ούτε διερμηνής ούτε αίθουσα. Γιατί είναι η μέρα που γίνονται όλες οι διαπραγματεύσεις και όλες οι αίθουσε είναι γεμάτες και όλες οι επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες συνεδριάζουν. Την Πέμπτη θα είναι πολύ αργά. Την Πέμπτη θα βρίσκαμε αίθουσα. Ναι, μπορεί να επιλέξει η Επιτροπή Πολιτισμού να κάνει μια έκτακτη συνεδρίαση. Στην περίπτωση όμως που δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, θα κάνουμε, θα το αναβάλουμε. Για ποιες τροπολογίες θέλετε να υποβάλουμε. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε με τους υπόλοιπους συντενιστές. Καταλαβαίνω την πρόταση της Προέδρου Καλό είναι που παρουσιάσαμε και τα τρία σενάρια. Για διάφορους λόγους, πολύ ειλικρινά, πιστεύω όπως είπε σε ένα πέτρα νωρίτερα, ότι σκόπιμο θα ήταν να περιμένουμε την ψηφοφορία ε, στην Ολομέλεια όσον αφορά την εντολή. Γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο περίπλοκη ήταν η κατάσταση. στο πλαίσιο της πρότασης ε, που ήταν το αντικείμενο δύσκολης ε, συζήτησης εντός της Επιτροπής μας και όλας ε, όλοι ήθελαν κάτι διαφορετικό οπότε θα έχουμε μεγάλη διαφοροποίηση στην ψηφοφορία νομίζω ότι θα βασιστεί και στις όποιες πολιτικές εξελίξεις τόσο όσον αφορά και άλλους συναδέλφους και άλλες επιτροπές ε, ε, όσο και βάσει όσο όσων θα γίνουν και στο Συμβούλιο. Έχω ακούσει ήδη τους συναδέλφους μας από την ομάδα που λένε να υποβάλουμε εκ των προτέρων κάποιες τροπολογίες εκ μέρους της Επιτροπής μας. Γι' αυτό θα έλεγα ε, για τη δεύτερη πρόταση που κάνεις και αφού πραγματοποιηθεί όλη η αντιπαράθεση που θα βασιστεί και σε περαιτέρω αξιολογήσεις και εντός της ομάδας μας ε, εκεί θα μπορέσουμε να διευρύνουμε τη συζήτηση να συμμετέχουν και άλλοι γιατί υπάρχουν πολλές και διαφορετικές απόψεις στην ομάδα μας για όλο αυτό. Ευχαριστώ. Ich sehe jetzt keine weiteren Wortmeldungen. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος το λόγο. Θα σας πω λοιπόν ότι ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα, την Πέμπτη, μπορούμε να συνεδριάσουμε στο Στρασβούργο. Το πρόβλημα είναι ότι στις 8 Ιανουαρίου, αν προσπαθήσουμε να βάλουμε συνεδρίαση, θα είναι τρία άτομα μες στην αίθουσα. Αυτό φοβάμαι. να προσπαθήσουμε, ζητώ συγγνώμη που το λόγο, να προσπαθήσουμε μετά την ψηφοφορία στο Στρασβούργο να έχουμε μιλήσει με όλους τους συναδέλφους από την Επιτροπή. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε και να βρούμε κάποια στιγμή μέσα στην εβδομάδα του Στρασβούργου. Πέμπτη πρωί κάποια στιγμή. Αλλιώς θα το κάνουμε στους συντονιστές. Έχω την εντύπωση ότι αν ε, κάνουμε επίσημα συνεδρίαση της Επιτροπής, ίσως είναι πιο δύσκολο, αλλά μέσω των συντονιστών. Κοιτάξτε, πρέπει να ληφθεί μια κανονική απόφαση όμως για αυτό το θέμα. Ποιες είναι οι τροπολογίες που θέλουμε να προωθήσουμε. Λοιπόν, οκ, θα προσπαθήσουμε για την επόμενη πέμπτη το πρωί να βρούμε κάποια στιγμή να συνεδριάσουμε. Δεν χρειάζεται μεγάλη συνεδρίαση. Θα συντονιστούμε και θα επικεντρώσουμε τη συζήτησή μας μόνο στο ποιε είναι αυτές οι τροπολογίες τη επιτροπή Πολιτισμού που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο κείμενο στην πρόταση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Η Γραμματεία ήδη, σα λέω, έχει επεξεργαστεί το θέμα. Έχουμε αναλυτικά την άποψή του Και με αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι μπορούμε να προετοιμαστούμε καλά έτσι ώστε την Πέμπτη το πρωί πολύ σύντομα σε μια σύντομη συνεδρίαση να συμφωνήσουμε γρήγορα. Εντάξει, συμφωνείτε. Ωραία. Περιμένουμε λοιπόν πρώτα την απόφαση της Ολομέλειας. Την τρίτη, την τρίτη. Ωραία. Οπότε να προχωρήσουμε στην ημερήσια διάταξη. Ψηφοφορίες. Σήμερα ψηφίζουμε την, το σχέδιο γνωμοδότησης Πρόκειται για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 20 η Έλγα Τρίπελ. Δεν είναι παρούσα, είναι εισηγήτρια, δυστυχώς δεν είναι σήμερα εδώ. 64 τροπολογίες, αρμόδια επί της ουσίας επιτροπής, είναι Επιτροπή Προϋπολογισμού. Αφού δεν είναι εδώ η συγγήτρια, μπορούμε λοιπόν να ψηφίσουμε κατευθείαν, δεν θα πάρει κανείς τον λόγο. Συμβιβαστική 1, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 16 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε το δεύτερο τμήμα, νομίζω απορρίπτεται, αρχή της ψηφοφορίας. Δεν δουλεύει. Για δοκιμάστε δίπλα. Πρέπει να ανάψει το πράσινο φωτάκι. Δουλεύει? Όχι. Να ξαναψηφίσουμε λοιπόν η δική σας ψήφος ξεχωριστά. Okay. Die Abstimmung ist geschlossen. Τέλος της ψηφοφορίας. Εννοείται ότι απορρίπτεται το δεύτερο σημείο με 15. Συμβαστική 4. Εποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, λέει η Πρόεδρο, αλλά δεν είναι σαφές. Συμβιβαστική 4 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, αρχή της ψηφοφορίας. 14 υπέρ, μία ψήφος κατά. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 Λάθος έκανα. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 40 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 41 υπέρ κατά αποχές νομίζω απορρίπτεται ψηφίζουμε όμως αρχή της ψηφοφορίας 41 τέλος εγκρίνεται η 41 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 46. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 και 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 49. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 50, α όχι η πέμπτη, λάθος, ε, 6 κατά αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 57. Α, όχι, όχι. Ελέγχουμε την 56. Τέλος. Απορρίφθηκε 56. Είχατε δίκιο. 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε το σύνολο του κειμένου αρχή της ψηφοφορίας τέλος Δεκατέσσερα υπέρ, Μία ψήφος κατά με μεγάλη πλειοψηφία λοιπόν εγκρίθηκε και συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Σαμπίνε. Η Σαμπίνε. Νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι ψήφισαν και πρέπει να φύγουν. Δεν είναι ότι δεν είναι ενδιαφέρουσα η συνεδρίαση, αλλά πρέπει να φύγουμε για να ψηφίσουμε σε μια άλλη επιτροπή. Δυστυχώς η Δευτέρα είναι μια μέρα με πολλές ψηφοφορίες. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στο θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης. Πρόκειται για την έκθεση Education and Train Monitor. Πρόκειται για μια ετήσια έκθεση, μια από τις πραγματικά για την ευαγγελματική κατάρτιση. Αναλύει την πρόοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με πολύ συγκεκριμένους στόχους ποσοτικούς στον τομέα αυτό της κατάρτισης. Σας παρακαλώ αν θέλετε να φύγετε, μην κάνετε θόρυβο. Πολύ συγκεκριμένα λοιπόν έχουμε πέντε κεντρικούς στόχους για το θέμα αυτό αφορά τη μείωση του ποσοστού αυτών που εγκαταλείπουν πολύ νωρίς το σχολείο, και βεβαίως ε, την βελτίωση των ποσοστών όσον αφορά αυτούς που εγκαταλείπουν το σχολείο με την ολοκλήρωση ενός πτυχίου, ενός κύκλου σπουδών, τη βελτίωση του επίπεδου στα μαθηματικά, στις επιστημονικές, ε, στους επιστημονικούς κλάδους, ε, ψηφιστική ιστορία, καλύτερη συμμετοχή επίσης των ενηλίκων σε σεμινάρια κατάρτισης και σε εκπαιδευτικούς ε, κύκλους. Ο κύριος Παγκόλσκι στην αρμόδια γενική διεύθυνση θα μας παρουσιάσει τα συγκεκριμένα αυτά αποτελέσματα, πολύ συγκεκριμένα και βεβαίως θα μπορεί να ακολουθήσει συζήτηση, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Έχετε το λόγο Έχετε 15 λεπτά. Μπορείτε όπως θέλετε βεβαίως να κατανέμετε μεταξύ σας οι δύο εκπρόσωποι της Γενικής Διεύθυνσης τον χρόνο ομιλίας αυτών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αυτή είναι η έκτη έκδοση της ε, ε, εκπαίδευσης της, του Education and Training Monitor. Ξέρετε, περιλαμβάνει δύο κομμάτια ε, ανάλυση αναχώρα με κάποια συστήματα επιδόσεων, καταμέτρηση επιδόσεων και το δύο, το δεύτερο κομμάτι περιλαμβάνει 28 κεφάλαια κατά χώρα. Ο συνάδελφός μου θα σα παρουσιάσει το κομμάτι αυτό της παρουσίασης. Το monitor αυτό παρουσιάστηκε από τον Επίτροπο Ναυράτσιτς ε, στις 9 Νοεμβρίου στις Βρυξέλλες. Όπως συνήθως ε, η δημοσίευση ακολουθεί μια συγκεκριμένη δομή. Κάνουμε αναθεώρηση των επιδόσεων των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε έξι εκπαιδευτικά ε, ε, σημεία αναφοράς. Εξετάζουμε τις διάφορους τομείς εκπαίδευσης και διαρευνούμε επίσης και τις εκπαιδευτικές δαπάνες των διαφόρων κρατών μελών Κάθε χρόνο έχουμε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. φέτο ε, εστιαζόμαστε στι ανισότητε. ένα σημαντικό θέμα δεδομένη της σημερινής κατάστασης στην Ευρώπη. Επιτρέψτε μου επίσης να προσθέσω ότι η φετινή έκδοση συνοδεύεται από πολλά νέα ηλεκτρονικά προϊόντα. Για πρώτη φορά η ηλεκτρονική δημοσίευση του monitor μπορείτε να το διαβάσετε σε Kindle και να έχετε ηλεκτρονική πρόσβαση στα δεδομένα υπάρχει ένα σύνολο βέλτιστων πρακτικών αλληλεπιδραστικοί χάρτες και διάφορα άλλα είναι μια μεγάλη προσπάθεια βελτίωσης της ε, ε, δημοσίευσης αυτής ώστε να γίνει πιο φιλική και για τους χρήστες μας τα κυρία μηνύματα Τη εκδοση αυτή ε, είναι τα εξή. Να σα. υπογραμμίσω πρώτα ότι βάσει του γενικού ε, στόχου η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να σημειώνει πολύ καλή πρόοδο. Όλε οι γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν μια, μια κατάσταση βελτιωμένη όσον αφορά την εγκατάλειψη, την πρώιμη εγκατάλειψη του σχολείου. Υπάρχουν διαφορές και μεταξύ χωρών και εντός των ίδιων χωρών. Εμείς ε, επισημαίνουμε τα απογοητευτικά αποτέλεσματα του τελευταίου γύρου της πίζας. Είναι ένα σημείο αναφορά που αφορά τους ανθρώπους με ελλειπείς επιδόσεις ε, σε τρεις τομείς ε, κατά βάση. Αντίθετα με τις προσδοκίες που υπήρχαν, η Ευρώπη φαίνεται να πηγαίνει προς τα πίσω. Ε, φαίνεται οι επιδόσεις των κρατών μελών να επιδενώνονται με εξαίρεση τρεις χώρες. Ειδικότερα όσον αφορά τις επιδόσεις στη ε, επιστημονικά μαθήματα, όπου φαίνεται να έχουμε πέσει από το στόχο από το 16% στο 20% ενώ ο στόχος ήταν 15%. Όσον αφορά τις επενδύσεις έχουμε αρχή, αργή αλλά σταθερή ανάκαμψη από τις περικοπές ε, ε, των δαπανών στην εκπαίδευση παρατηρείται τώρα ελαφριά αύξηση. Και πάλι βάσει των ε, στοιχείων που έχουμε οι ανισότητες παραμένουν στην Ευρώπη. Τα εκπαιδευτικά συστήματα έχουν αναπτύξει μηχανισμούς για να είναι λιγότεροι οι αποκλεισμοί και πιο ε, μεγάλες επιδόσεις, ωστόσο τα πράγματα παραμένουν ε, δύσκολα. Όσον αφορά τις συνέπειες των ανισοτήτων ε, στον επαγγελματικό τομέα και στις σχετικές πρόπτικες εκεί, είναι σαφές ότι τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα. Οι μαθητές και οι μαθήτρες που φεύγουν στα πρώτα χρόνια της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το σχολείο ε, τείνουν να παραμένουν άνεργοι. Το 44% των ε, ε, ανθρώπων 18 έως 24 ετών μόνο εργάζονταν το 2016. Αν δείτε ολόκληρο το φάσμα σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς όσον αφορά την ανεργία όσοι δεν έχουν, έχουν μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση το 16,6% μόνο ε, ε, είναι απασχολημένοι. Υπάρχει επίσης ένα σαφής κίνδυνος ε, μετάβαση στη φτώχεια ή στον κοινωνικό αποκλεισμό. Να επιστήσω την προσοχή σας στη διαφάνεια που μιλάει για τα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης όσον αφορά τις ανισότητες εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με τη χώρα. Προφανώς το ζήτημα της ένταξης των μεταναστών ε, επηρεάζει σημαντικά την κατάσταση σε πολλές χώρες. Τα άτομα που εξετάζει η πίζα έχουν αυξηθεί κατά 22,5 ε, ποσοστίες ε, μονάδες ορισμένες χώρες. Ε, μιλάμε για μετανάστες πρώτης γενιάς. Τώρα, σε σχέση με, τον, με το κοινωνικό υπόβαθρο, και αυτό παίζει μεγάλο ρόλο στις χαμηλές επιδόσεις μαζί με την εκπαίδευση με την παιδεία των γονιών όσον αφορά το φύλλο τώρα ε, ε, στις γυναίκες, οι γυναίκες ε, μορφώνονται καλύτερα ενώ έχουν χαμηλότερες επιδόσεις όσον αφορά τις ευκαιρίες για απασχόληση και για παιδεία. Σε αυτήν εδώ τη διαφάνεια βλέπετε μια εικόνα για όλη την Ευρώπη. Το χάσμα του φύλου στον τομέα της εκπαίδευσης είναι σχεδόν 10% και όσον αφορά την απασχόληση περίπου έχουμε το ίδιο ποσοστό, την ίδια διαφορά μεταξύ φύλων. Όσον αφορά τα άτομα χαμηλών επιδόσεων βλέπετε εδώ και αυτό που ανέφερα πρωτήτερα ε, διαφορά μεταξύ χωρών και μεταξύ κοινωνικών ομάδων, ειδικότερα των μειονεκτουσών ε, ομάδων ε, από χαμηλό κοινωνικό υπόβαθρο, είναι πιο ευάλωτε αυτέ οι ομάδε σε σχέση με αυτού που έρχονται από τα ανώτερα κλιμάκια του οικονομικού υπόβαθρου. Όσον αφορά του μετανάστε και πάλι το ζήτημα αυτό ε, εδώ βλέπουμε πολύ και σαφώς τα πράγματα όσον αφορά ε, τους, ε, τα άτομα χαμηλών επιδόσεων και εδώ βλέπετε ότι οι διαφορές είναι πολύ σημαντικές μεταξύ των μη μεταναστών και των τοπικών πληθυσμών. Έχουμε προετοιμάσει φύλλα εδώ με όλες τις ε, διαφάνειες. Δεν θα σας πω, δεν σας αναφέρω τα πάντα, όλα τα σημεία αναφοράς, αλλά να σας πω ότι όσον αφορά τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, η Ευρώπη εξακολουθεί να φέρνει περίπου το 5% του ΑΕΠ, αλλά υπάρχουν τεράστιες διαφορές ακόμη μεταξύ των κρατών μελών. Να σας παραπέμψω στα λεπτόμερη ε, δεδομένα, θα σας παραπέμψω που υπάρχουν αφού υπάρχει περιορισμένος χρόνος και θα δώσω το λόγο στον συναδελφό μου που θα σας παρουσιάσει το δεύτερο κομμάτι του δημοσιεύματος. Is working? Yes. Uh, thank you, thank you, Madam Chair, for Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, για την δυνατότητα που μου δίνετε. Είδα ότι έχουν μοιραστεί στους συναδέλφους σας αντίγραφα ε, της ε, έκθεσης. Did you look further at the points which Jan has, has, has elaborated here? Ε, έχουμε λοιπόν διάφορα στοιχεία, ε, ε, αλλά αυτό που θα ήθελα να αναφερθώ εδώ, ακριβώς επειδή ενδιαφέρεστε πάρα πολύ στις, στην έλλειψη ισότητας, πρέπει να πούμε ότι αυτή η έλλειψη ισότητας υπάρχει ακόμα, επιμένει και μάλιστα σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις 28 χώρες μέλη γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό της έλλειψης ισότητας. Ωστόσο, μιλάμε εδώ για διαφορετικές προσεγγίσεις, για διαφορετικά υπόβαθρα και, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα εξακολουθεί να παραμένει. Ε, στο δεύτερο τόμο βλέπετε και κάποια καλά παραδείγματα ε, για πόλεις, ε, περιφέρειες, οι οποίες μπορεί να βρίσκονται και στην ίδια ε, χώρα. Εν πάση περιπτώσει, για να επανέλθω σε κάποια από τα σημεία που ανέφερε ο συνάδελφός μου, να πω τα εξή. Έχουμε την αίσθηση ότι οι χώρες οι οποίες έχουν ήδη δώσει, έχουν ήδη τα αποτελέσματα για την πίζα, ότι εξακολουθούν οι ίδιες χώρες να έχουν υψηλά αποτελέσματα και επιδόσεις όπως η Φιλανδία ας πούμε. Ε, οι χώρες οι οποίες ε, είναι χώρες καλών αποτελεσμάτων επιδόσεων και αριστείας ε, είναι αυτές οι οποίες έχουν και μικρότερη διάσταση όσον αφορά το θέμα της ισότητας. Και τα τεκμήρια της έρευνάς μας καταδεικνύουν ότι υπάρχουν οι ίδιες διαπιστώσεις ε, σε αυτές τις χώρες με τις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλά αποτελέσματα και το κυριότερο στοιχείο που έχουν κοινό είναι ότι είναι χώρες οι οποίες παρουσιάζουν πολύ μεγάλες διαστάσεις ε, όσον αφορά ε, τα αποτελέσματα. Ας πούμε διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών και όσον αφορά την ισότητα και όσον αφορά την ισομερή πρόσβαση στην εκπαίδευση. Για 15 χρόνια λοιπόν στην Πίζα βλέπουμε ότι οι διαστάσει εκεί μπορεί να είναι στην ίδια, σε ορισμένε χώρες, στην ίδια χώρα, ανάλογα την περιφέρεια, μπορεί να είναι λέω πάρα πολύ μεγάλες. Ε, αυξάνει ο αριθμός των χωρών οι οποίες έχουν ε, ε, ε, μη ικανοποιητικά αποτελέσματα. Επίσης ε, γίνεται μια προσπάθεια να ακολουθήσουμε τα στοιχεία και στον πρώτο και στο δεύτερο τόμο όσον αφορά την ε, ε, ολοκλήρωση των σπουδών, της διαδικασίας μάθησης, τη μη κατάληψη του σχολείου, την συνέχιση των σπουδών κτλ. Επίσης έχουμε δει όσον αφορά την απορρόφηση της χρηματοδότησης. Βλέπουμε ότι υπάρχει δυνατότητα μεγαλύτερης απορρόφησης. Έχουμε φτάσει στα επίπεδα προκρίσης. Σε ένα τρίτο των χωρών ε, μελών δεν έχει όμως ανακάμψει ε, η δαπάνη για την εκπαίδευση. Στα δύο τρίτα έχουμε φτάσει, όπως είπα και προηγουμένως, στα επίπεδα πριν από την κρίση. Ε, όσον αφορά τώρα την μαθητεία, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα. Έχουμε επιμείνει στο σημείο αυτό και ε, αυτό το στοιχείο της μαθητείας του vocational training δηλαδή ε, έχει προωθηθεί πάρα πολύ σε ορισμένες ε, χώρες. Είναι πολύ, όλο και περισσότεροι πλέον αυτοί οι οποίοι αποφασίζουν να ακολουθήσουν αυτήν την οδό της μαθητείας και ε, ε, σε αυτού του είδους τη μαθητεία βλέπουμε ότι ε, προσανατολίζονται πολλοί νέοι με χαμηλές επιδόσεις και επομένως βλέπουμε ότι από τις χαμηλές οικονομικές και κοινωνικές ομάδες τελικά οι περισσότεροι στρέφονται προς την μαθητεία έτσι ώστε να αποκτήσουν κάποια βασικά προσόντα. Λοιπόν, κυρία Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτά ήθελα να σας πω. Σας ζητώ όλους, από όλους, να δείτε προσεκτικά αυτούς τους δύο τόμους να δείτε κυρίως ε, την ε, σχέση ανάμεσα στις επιδόσεις ε, και τα σημεία αναφορά στα benchmark τα οποία έχουμε μελετήσει. Υπάρχουν, επίσης σας καλώ να δείτε τα ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία έχουν προκύψει από την ανάλυση αυτή ε, έχουμε σημαντικές εξελίξεις και ενδιαφέρουσες και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Θα ήθελα να τα δείτε αυτά γιατί έχουμε περιλάβει και κάποια ε, παραδείγματα και εν πάση περιπτώσει σας ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να παρουσιάσουμε την έκθεση αυτή. Πάρα πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Θερμά σας ευχαριστώ για την προετοιμασία αυτής της έκθεσης. Πραγματικά διαπιστώνουμε πράγματα που τα υποψιαζόμασταν. Εννοείται ότι η καλή εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει στα πρώτα πρώτα χρόνια της ηλικίας. Το κλειδί είναι βεβαίως να συνεχίσει αυτή η καλή πρώτη εκπαίδευση και στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στο πανεπιστήμιο. Είναι καθοριστική λοιπόν αυτή η έκθεση για την περαιτέρω δική μας εργασία και πιστεύω ότι πραγματικά οι δύο συνάδελφοι από την Επιτροπή μας παρουσίασαν εδώ με πολύ λεπτομερή τρόπο τις διαφορές που συνεχίζουν να υπάρχουν, παραδείγματο χάρη μεταξύ των ε, δύο φίλων, τα κορίτσια έχουν εξαιρετικά αποτελέσματα το σχολείο, στις σπουδέ, όμως κατόπιν καθυστερούν στη σταδιοδρομία τους και τα αγόρια τα ξεπερνούν. Είναι βεβαίως πολύ σημαντικό το θέμα αυτό της επαγγελματικής ε, κατάρτισης, της επαγγελματικής ε, σταδιοδρομίας, πως ε, υπάρχει συνάρτηση μεταξύ των σπουδών και της συνέχειας είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι το πτυχίο, το πανεπιστημιακό, όσο σημαντικό και αν είναι, θα πρέπει να ανοίγει τις πόρτες σε μια επαγγελματική σταδιοδρομία. Όποιο και να είναι αυτό, επαναλαμβάνω θα πρέπει να υπάρχει η ίδια αξία και η ίδια δυνατότητα να ενσωματωθεί κάποιος στην αγορά της εργασίας, όποιο και να είναι το πανεπιστήμιο, όποιο και να είναι η σχολή, έτσι ώστε να μην υπάρχουν λιγότερο σημαντικά ή περισσότερο σημαντικά πτυχία, είτε πρόκειται για επαγγελματική κατάρτιση, είτε πρόκειται για ακαδημαϊκές σπουδές, δεν χρειαζόμαστε μόνο αρχιτόκτονες και γιατρούς. Χρειαζόμαστε και ανθρώπους οι οποίοι τελικά να χτίζουν αυτά τα σπίτια. Να υλοποιούν τα σχέδια τα αρχιτεκτονικά. Και βεβαίως είναι πάρα πάρα πολύ λυπηρό να βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης σε πολλά κράτη δεν επενδύουν πλέον οι αρχές στην εκπαίδευση, στο εκπαιδευτικό σύστημα και ότι υποχωρεί η προσπάθεια για καλύτερη εκπαίδευση. Μας εγκατέλειψαν κάποιοι συνάδελφοι γιατί έπρεπε να ψηφίσουν σε άλλες επιτροπές, αλλά κάποιοι είναι εδώ και φυσικά θα δώσω αμέσως το λόγο στον κύριο Στογεύσκη. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την ε, Επιτροπή για όλα αυτά τα αποτελέσματα. Ωραίο είναι που έχουμε ένα έγγραφο τόσο γεμάτο πληροφορίες ε, τέτοιες ποιότητας. Θα είχα να κάνω περισσότερες ερωτήσεις αν μου είχαν έρθει τα αυτά πιο νωρίς. Ε, να προσθέσω και αυτό το σχόλιο στα σχόλιά μου, οπότε θα περιοριστώ σε λίγα. Ε, κύριε Πακούσκη, πολύ συχνά οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν τη διάκριση μεταξύ του εικονικού και του πραγματικού κόσμου, μεταξύ της αλήθειας ε, και του ψεύδους. Ακόμη και οι ενήλικες δυσκολεύονται με το ίδιο πράγμα. Αυτό το σημείο το λαμβάνεται υπόψη ε, όταν σχεδιάζουμε την εκπαίδευση και τον εκπαιδευτικό κόσμο ε, καθορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι ε, συγκεκριμένες εργασίες ώστε να μαθαίνουν ε, οι νέοι να διακρίνουν την προπαγάνδα από την πραγματικότητα, το ψέμα από την αλήθεια, να κάνουν τη διάκριση μεταξύ του πραγματικού και του ε, φανταστικού κόσμου. Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με την ακρόαση της Πέμπτης. Θα συζητήσουμε για τη συλλήψη της παιδείας. Ξέρουμε ότι αυτή η ακρόαση, αυτός ο αποκλεισμός αφορά τους μετανάστες, τους ανθρώπους με αναπηρίες σε κάποιο επίπεδο. Ήθελα να μου πείτε κατά πόσο ο αποκλεισμός αυτός οφείλεται και σε ελλείψεις της παιδείας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο ζήτημα το οποίο εφήγει είναι πάρα πολύ σημαντικό. International community, not uh, Europe alone. Um, there are several... Υπάρχουν πάντως ε, αρκετά εργαλεία, είτε που υφίστανται ήδη, είτε που είναι υποσυζήτηση. Η συζήτηση ε, η Κομισιόν συγγνώμη, έχει συγχρηματοδοτήσει κάποιες προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα ε, κράτη-μέλη ε, να αναπτύξουν τις πολιτιακές ικανότητες στους νέους και επίσης να αναπτύξουν την ικανότητα που έχουν να ε, αντιμετωπίσουν πράγματα της καθημερινότητας ε, βγάζοντάς τους κατά κάποιο τρόπο από τον ηλεκτρονικό κόσμο στον οποίο έχουν μάθει να ζουν. Ένα από τα εργαλεία τα οποία έχουμε χρησιμοποιήσει και μάλιστα τώρα έχουμε και διαθέσιμα ε, τα αποτελέσματα και σκεφτόμαστε να τα βάλουμε και στο τώρα ακριβώς αφορούν αυτό το θέμα. Επίσης ε, ε, γίνονται συζητήσεις όσον αφορά ε, τον επόμενο γύρο της πίζα το 21-24 και εκεί θα βάλουμε τις λεγόμενες global competencies έτσι ώστε να μπορέσουμε να μετρήσουμε με αποτελεσματικό τρόπο την ικανότητα των νέων να λειτουργήσουν ε, σε αυτό το ε, περιβάλλον ε, στο οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν πραγματικά περιστατικά και στοιχεία γιατί απομακρύνονται καμιά φορά από αυτόν τον πραγματικό κόσμο ακριβώς λόγω της χρήσης πολλών ηλεκτρονικών συσκευών. Και επομένως θέλουμε να μετρήσουμε την πραγματική τους ικανότητα να κινηθούν στον πραγματικό κόσμο. Κοιτάξτε, ε, όσον αφορά το άλλο θέμα, ναι, βεβαίω ε, το γνωρίζουμε και το θέλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Το θέμα του αποκλεισμού από όψη πολιτιστική είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το είπατε κι εσείς έχει προκύψει το θέμα αυτό κυρίως σε σχέση με την ένταξη ε, και συμπερίληψη στην κοινωνία των μεταναστών και η χρήση ε, των ε, εργαλείων του, πολιτισμού και της εκπαίδευσης ε, για την ενδυνάμωση της αίσθησης του ανήκειν ε, είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το αναγνωρίζουν όλοι και επομένως είναι πραγματικά πρόθεσή μας να υποστηρίξουμε τις διαδικασίες αυτές. Και σε σχέση με το δεύτερο ερώτημα ε, πραγματικά έχω την ίδια απάντηση με τον συνάδελφό μου. Ε, δεν έχω κάποιο παράδειγμα αποκλεισμού από τα πολιτιστικά αγαθά κάποιων ε, νέων. Πάντως, αν δείτε ας πούμε για το Βέλγιο, στην Φλάνδρα, υπάρχουν νέες ε, πρακτικές ε, οι οποίες αφορούν ακριβώς την ενδυνάμωση της δυνατότητας των νέων να αντιμετωπίσουν ε, την πραγματική ζωή και για να αποκτήσουν τέλος πάντων νέες δεξιότητες. Τα υπόλοιπα συμφωνώ ότι μπορούμε να τα περιλάβουμε και στο monitor την επόμενη φορά. Ευχαριστώ. το θέμα των ψηφιακών ε, δεξιοτήτων κατά πόσο στα κράτη-μέλη το θέμα που αφορά τα μέσα, το θέμα που αφορά την ψυχιακή τεχνολογία έχουν ενσωματωθεί στα διάφορα εκπαιδευτικά συστήματα, τα προγράμματα, πόσο υποστηρίζονται δηλαδή. Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να το εξετάσουμε για το μέλλον, να βρούμε συγκρίσιμα αποτελέσματα, να μετρήσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέρον για μας. Θέλουμε συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία, γιατί ξέρουμε επίσης ότι αυτές οι δεξιότητες είναι καθοριστικές και σίγουρα θα επηρεάζουν την επαγγελματική ζωή των νέων ε, Ευρωπαίων. Επίσης, τα θέματα του πολιτισμού, πολιτιστικά θέματα, κατά πόσο στα κράτη-μέλη, στη σχολική εκπαίδευση αλλά και στην επαγγελματική κατάρτιση, ο πολιτισμός παίζει ένα ρόλο. Ποια είναι η επίπτωση αυτών των δεξιοτήτων όταν υπάρχουν οι λεγόμενες soft skills. Πώς επηρεάζουν δηλαδή την ενσωμάτωση αυτών των συγκεκριμένων ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Μπορείτε να μας πείτε αν αυτό μπορεί να συμπεριληφθεί σε μια μελλοντική σας έκθεση. Δεν βλέπω όμως ερωτήσεις από την αίθουσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο που ήρθατε σήμερα εδώ, που μας κάνατε αυτή την παρουσίαση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη την προσπάθεια που βάλατε σε αυτήν την έκθεση. Είναι πολύ σημαντική η πληροφόρηση για μας, για την Επιτροπή μας. Γιατί αυτό που είναι ενδιαφέρον να κοιτάξει κανείς τι συμβαίνει και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στη δικιά του. Ποιε είναι οι καλές πρακτικές, τα επιτυχή σενάρια, τι μπορεί να βελτιωθεί στο καθενός ε, τη χώρα αν υιοθετήσουμε κάποιες άλλες ε, πρακτικές, κάποιες άλλες ιδέες, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια πραγματικά επιτυχημένη ευρωπαϊκή παιδεία, ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να έχει τα επιθυμητά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως και τους δυο σας για αυτή την έκθεση και αν λάβετε υπόψη και τις παρατηρήσεις μας θα σας είμαστε ευγνώμονες. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Πρόκειται για τη γνωμοδότηση που πρέπει να εξετάσουμε, σχέδιο γνωμοδότησης. Πρόκειται για τον προϋπολογισμό για το 2016. Ο συνάδελφος το Γεύσκι είναι εισηγητής. Η 7η Δεκεμβρίου στις 4 είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στις 23 Ιανουαρίου εδώ στην Επιτροπή. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, 8 Δεκεμβρίου στις 4. 23 Ιανουαρίου θα ψηφίσουμε. και το Μάρτιο του 2018 θα ψηφίσει η ε, επί αρμόδια επιτροπή, η Επιτροπή Προϋπολογισμού. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε για την διόρθωση που μόλις κάνατε. Ε, γιατί η 8η Δεκεμβρίου είναι πολύ κοντά. Να υπενθυμίσω πάντως ότι οι προτάσεις μας ε, έχουν σημαντική επίπτωση στους μελλοντικούς προϋπολογισμούς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να υποβάλουμε τροπολογίες οι οποίες ε, θα επηρεάσουν μελλοντικούς σχεδιασμούς και θα αποτελέσουν ε, και έναν τρόπο υπολογισμού των εκτιμήσεων τέλο πάντων της Επιτροπής Προϋπολογισμού. Να σας πω ότι μπορώ να είμαι ήπια ικανοποιημένος και για ποιο λόγο λόγο γιατί η ε, χρηματοδότηση προγραμμάτων όπως ας πούμε η Δημιουργική Ευρώπη, Creative Europe ή η Ευρώπη για τους ε, πολίτες. Ε, πώς να σας το πω, είναι προγράμματα ε, τα οποία έχουν χαμηλή εκτέλεση και βεβαίως είχαν και χαμηλή χρηματοδότηση. Γνωρίζουμε ότι και παραδοσιακά το ποσοστό επιτυχίας των προγραμμάτων ήταν 16 και 11% αντιστοίχους. Όσον αφορά τώρα, αντιστοίχως, όσον αφορά τώρα την ε, διαφοροποίηση των ε, πληρωμών, να σας πω ότι ε, οποτεδήποτε είναι δυνατόν θα πρέπει να μιλάμε για το Erasmus Plus, ε, να μιλάμε για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, να μιλάμε για την ε, δανειοδότηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί εάν θέλουμε οι δικαιούχοι μέχρι το 2020 να είναι 4 εκατομμύρια θα πρέπει να είναι επαρκής και ο μηχανισμός χρηματοδότησης. Ευχαριστώ. Ο κύριος... Ο κύριος Λουτζιμόγκανο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι έχουν τα πράγματα και πρέπει να κινηθούμε αντιστοίχως. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο τον συνάδελφο Σδρογεύσκη να τον ευχαριστήσω για το σχέδιο γραμμοδότησης το οποίο υπέβαλε, το οποίο κατά την άποψή μου παρουσιάζει σειρά στοιχείων που ε, μπορούμε, ε, με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά ε, τον προϋπολογισμό του 2016. Συμφωνώ μαζί του ότι θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε να δείξουμε ποιε είναι οι ανάγκες της Επιτροπής μας για το μέλλον. Ε, εγώ θα υπογραμμίσω ορισμένα στοιχεία. Πρώτον, στην έκθεση του ελληνικού συνεδρίου όσον αφορά ε, τα σοβαρά ε, σφάλματα, τα προγράμματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Πολιτισμού δεν αναφέρονται ποτέ, τουλάχιστον όχι ρητά. Πράγμα που με οδηγεί στο συμπέρασμα ότι από άποψη λογιστική η εργασία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι σωστή και επενετέα. Δεύτερον, ε, σύμφωνα με τις ε, διαδικασίες ε, απαλλαγής πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν κάποια ζητήματα. Δηλαδή, ε, η δικιά μας ε, εντολή ως ε, βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιλαμβάνει και τον δημοκρατικό έλεγχο της πραγματικής υλοποίησης των ευρωπαϊκών πολιτικών στα κράτη-μέλη και δέσμευσή μας επί τη βάση του λογιστικού ελέγχου του ελεγκτικού συνεδρίου είναι να ελέγξουμε εάν οι πόροι οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν και μέσω των δικαιούχων έχουν καλύψει τους στόχους για τους οποίους είχαν αρχικά δοθεί. Κατά αυτή την έννοια θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε ότι σημαντικά ποσοστά λάθους ε, αναφέρονται και φέτος όπως και άλλες χρονιές σε μία σα τομέων ε, στους ε, οποίους υπάρχει μεικτή αρμοδιότητα μεταξύ κρατών μελών και ευρωπαϊκών Ένωσης. Ε, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον για τους νέους στον Έρασμο Πλάς ε, υπάρχουν κάποια ζητήματα και επίσης ε, θα πρέπει οι δικαιούχοι να ε, ε, ε, συμπεριληφθούν περισσότερο ε, σε έναν υποπρογραμματισμό του προγράμματος. Το λέω αυτό γιατί πρόκειται για θέση του Κοινοβουλίου που έχει μάλιστα δηλωθεί και υπερψηφιστεί σε πολλές εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να το επαναλάβουμε λοιπόν. Επίσης, όπως σωστά υπογράμμισε και ο εισηγητής, ε, τα ε, χαμηλά ποσοστά επιτυχίας για την Ευρώπη, για τους πολίτες και τη δημιουργική Ευρώπη καταδεικνύουν σαφώς ε, και αυτό θα πρέπει να μας ε, βοηθήσει και στο επόμενο MFF ε, καταδεικνύει λέω τις οικονομικές ανάγκες χρηματοδοτικές ανάγκες αυτών των προγραμμάτων. Επίσης όσον αφορά τον εκτελεστικό οργανισμό εκπαίδευση του και πολιτισμού ο μηχανισμός εγγυήσεων για τον ε, τομέα του πολιτισμού ε, έχει ε, χρησιμοποιηθεί μονάχα για δύο υπηρεσίες. Επίσης, ορίζεται ως ένα πρόγραμμα το οποίο μονάχα στο τρίτο χρόνο εκτέλεσης έχει φτάσει σε ένα επίπεδο οριμότητας. Αναφέρομαι, αναρωτιέμαι λοιπόν, εάν, και στρέφουμε και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν ε, ε, αν πρέπει κάθε φορά να ξεκινάμε από το μηδέν ε, για κάθε πρόγραμμα ή μήπως θα έπρεπε να διατηρήσουμε τις δομές αυτές οι οποίες έχουν αποδείξει ότι λειτουργούν καλά. Και εκεί, από εκεί και πέρα να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία. Παραμένει βεβαίως και ένα άλλο οριζόντιο πρόγραμμα ουσίας. Το 2016 είχαμε ε, ε, ένα ρεκόρ ε, πληρωμών που μετατέθηκαν για, επόμενους, για επόμενες λογιστικές χρονιές. Πιστεύουμε ότι εδώ θα πρέπει να προσέξουμε και θα πρέπει να υπάρχει και προϋπόθεση, δηλαδή ότι κάθε χρόνο να υπάρχουν απαραίτητες προμήθειες για τους πόρους πληρωμής έτσι ώστε να μην υποχρεώνονται οι χώρες να μειώνουν τον προϋπολογισμό που ε, προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα το οποίο δεν μπορεί να μας βρει σύμφωνο στη δικιά μας Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ποιος δεν θέλει να πάρει το λόγο. Κανείς. Κύριε Στρογεύσκη, θέλετε πάλι το λόγο. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και τον συνάδελφο Μόργανο για την παρέμβασή του, με την οποία συμφωνώ 100%. Αναφέρθηκε ότι η Επιτροπή ε, Πολιτισμού δεν λαμβάνεται υπόψη ε, με ε, τις δικές της δαπάνες και ανάγκες. Αυτό είναι θέμα του προϋπολογισμού αλλά και κοινή πρακτική. Η πρακτική αυτή μεταφράζεται ε, σε πάρα πολύ μικρό, για να μην πω άνευ σημασία, τμήμα του προεπολογισμού για την δικιά μας Επιτροπή. Έχετε δίκιο κύριε Μόργαν όταν λέτε ότι εμείς έχουμε μεγάλη ευθύνη για τον έλεγχο ε, το, της εκτέλεσης του προπολογισμού κατά τη διάρκεια του έτους δεν ε, μας ενδιαφέρει μονάχα η ποσότητα ε, των χρημάτων και των πόρων αλλά και ε, η ποιότητα. η Ευρώπη για τους πολίτες και η Δημιουργική Ευρώπη είναι δύο εξαιρετικά προγράμματα τα οποία θα πρέπει να συνεχίσουν και μάλιστα να ενισχυθούν. Πολύ σωστές είναι οι παρατηρήσεις του συναδέλφου λοιπόν και εγώ θα ήθελα να κάνω μία ακόμη παρατήρηση την οποία ξεχάσαμε και ο υποφαινόμενος και ο συνάδελφος θα πρέπει να δούμε τα πιλωτικά προγράμματα, να τα χρησιμοποιήσουμε, να τα εκμεταλλευτούμε και να δούμε βάσει των πιλωτικών προγραμμάτων ποια είναι τα προγράμματα τα οποία μπορούν καλύτερα και να υλοποιηθούν και με καλύτερα αποτελέσματα και επί τη βάση αυτών να βρούμε νέες ε, καινοτομίες έτσι ώστε να μην περιορίζεται η δραστηριότητά μας ε, και να μην γίνονται άκαμπτες ε, οι προτεραιότητά μας και βεβαίω ε, να μειωθεί η διαφορά ανάμεσα σε υποχρεώσει και πληρωμές, το είπα και προηγουμένω αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πληρωμές, υποχρεώσει. Κάθε χρόνο έχουμε τις ίδιες συζητήσεις και δυσκολίες εάν δεν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε εγκαίρως. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Στογεύσκη. Λοιπόν, κύριε Μόργανο, Νομίζω ότι θα συνεργαστείτε με εξαιρετικό τρόπο. Είμαι σίγουρη ότι η έκθεση για την απαλλαγή θα είναι έτοιμη εγκαίρω και τέλος Ιανουαρίου θα μπορέσουμε να την ψηφίσουμε. Περνάω στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Κύριε Στογεύσκη, πάλι εσείς είστε ο εισηγητής. Πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας που αφορά τους διαρθρωτικούς αυτούς ε, τις ε, διαρθωτικές αυτές και οικονομικές ε, δυσκολίες και εμπόδια όσον αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό. Σχέδιο έκθεσης θα υποβληθεί 21-22 Φεβρουαρίου και η ε, υποβολή των τροπολογιών στις 28 Φεβρουαρίου. Θα ψηφίσουμε τον Απρίλιο. Ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας σας. Ε, ε κοινή απόφαση ήταν να, να ε, ξεχωρίσουμε, να διαχωρίσουμε το κέντρο μεταφράσεων. Χάρη σε αυτό μπορέσαμε να διοργανώσουμε μία ακρόαση εδώ στην Επιτροπή μας ώστε να συζητήσουμε το θέμα αυτό. Τι είπαμε λοιπόν, πρέπει πρώτα απ' όλα να ενισχύσουμε το θεσμό αυτόν. Αλλά είπαμε επίσης ότι και οι δημοσιονομικές περικοπές για το μεταφραστικό κέντρο δεν είναι αιτιολογημένες. Αυξάνεται ο ρυθμός των πελατών, αυξάνονται τα αιτήματα μετάφρασης ε, αυξάνονται τα χρήματα που απαιτούνται και οι αμοιβέ και ήταν πολύ περίεργη αυτή η περικοπή που ζήτησαν. Εντάξει, ήταν μόλι 5% αλλά η Επιτροπή εφιστά την προσοχή μας στο γεγονό ότι οι μειώσει αυτές, οι περικόπες αυτές ε, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν ε, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να ενσωματωθεί και να ενδυναμωθεί ο θεσμός. Οπότε, εν συντομία, χαίρομαι που έχει υπάρξει αυτή η έκθεση για τον σε σχέση με τον προπολογισμό. Σας ευχαριστώ. Εγώ ήμουν στο άλλο θέμα. Εσείς μιλήσατε για το κέντρο μετάφραση. Εγώ μιλούσα για τα εμπόδια στην πρόσβαση στον πολιτισμό. Εν πάση περιπτώσει, δεν πειράζει, μιλήσουμε για το κέντρο μετάφρασης. Ευχαριστώ. Επειδή όπως είπατε και εσείς ε, Πρόεδρε είναι σημαντικό το θέμα αυτό. Ε, είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν ε, γιατί είπαμε ότι έπρεπε να κοιτάξουμε από πιο κοντά το ζήτημα αυτό. Όπως ξέρουμε το ελεκτικό συνέδριο είπε εδώ ότι πρέπει να έχουμε χρηστή διαχείριση και ισότιμη διαχείριση. Το κέντρο αυτό είναι υπευθύνο για τις μεταφράσεις σε όλες τις γλώσσες για όλα τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί το λέω αυτό, διότι επιφορτίζεται για μεταφράσεις για τους άλλους οργανισμούς ε, πελάτες που πρέπει να πληρώνουν το κέντρο για αυτές τις υπηρεσίες. Ε, ε, από αυτό, αυτά είναι τα κονδύλια ουσιαστικά, εκεί πάνε τα κονδύλια. Αλλά εδώ υπάρχει ένα άλλο στοιχείο ότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι οι οργανισμοί να χρησιμοποιούν το κέντρο. Ενίοτε χρησιμοποιούν ε, εσωτερικές υπηρεσίε μετάφρασης. Κάτι που οδηγεί σε διπλασιασμό των συστημάτων. Επικάλυπτο. Αλλά φυσικά θα πρέπει αυτό να το δούμε και σε συνδυασμό και με μια άλλη πτυχή που είναι η πτυχή της ποιότητας. Κάτι άλλο που δεν αναφέρθηκε, αλλά θα μπορούσαμε να το σκεφτούμε με τον κύριο Στρογεύσκη, αν χρειάζεται να το αναπτύξουμε περαιτέρω, ε, αυτό το θέμα. Οι υπηρεσίε τιμολογούνται, ε, πρέπει να τιμολογούνται με τρόπο λογικό. Ταυτόχρονα πρέπει να ε, ορίζονται σε συνεργασία με αυτούς που ζητούν τις υπηρεσίες. Μετά είπε, όπως είπε ο συναδέλφος, υπήρξαν σοβαρές περικοπές και ε, υποχρεώθηκε το κέντρο να μειώσει και το προσωπικό κατά 5%. Κατά την άποψή μου, λοιπόν, πρέπει να διασφαλίσουμε την ποιότητα των μεταφράσεων σε όλες τις γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ εξάλλου με τον ε, εισηγητή. Δεν θα επιθυμούσαμε μελλοντικές περικοπές ε, στον προϋπολογισμό και στο προσωπικό συμφωνώ με τον συνάδελφο Στρογεύσκη, πρέπει να δεσμευτούμε για την ποιότητα και θα πρέπει να μας απασχολήσει περαιτέρω το ζήτημα των εσωτερικών διαγωνισμών και τα αποτελέσματά τους, διότι τα αποτελέσματά τους δεν είναι πάντα ικανοποιητικά. Από αυτή την άποψη λοιπόν ε, να συμφωνήσω με την έκκληση που υπάρχει στο κείμενο όσον αφορά την πολύ ευαίσθητη πτυχή της ε, εκπαίδευσης, ε, της κατάρτισης των απαραίτητων ικανοτήτων για να πραγματοποιεί κανείς ε, τη μετάφραση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Κύριε Στογεύσκη, θέλετε να επανέλθετε στο σημείο αυτό. Ναι, είναι προφανές ότι εδώ μιλάμε για τις γραπτές μεταφράσεις. Είναι γεγονός ε, ότι έχουμε ένα ψηλό ποσοστό ε, όσον ε, αφορά τις δυνατότητες εσόδων και πόρων για να καλύψουμε αυτές τις δυνατότητες μετάφρασης. Συγχαίρουμε λοιπόν το κέντρο για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τους πόρους. Απ' την άλλη μεριά βεβαίως και αφού τους έχουμε σύγχαρου, ρί θα πρέπει να δούμε ε, και το πώς μπορεί να επιτευχθεί η σωστή μετάφραση. Θα πρέπει να σταματήσουν οι περικοπές, θα πρέπει ε, να σταματήσουν, ε, θα πρέπει να, να δοθεί η δυνατότητα να δουλέψουν καλά οι μεταφραστές αυτού του κέντρου. Ευχαριστώ. 8 Δεκεμβρίου στις 4 είναι η προθεσμία για την υποβολή των τροπολογιών. Περνάμε στο σημείο 7 της ημερήσιες διάταξης, αυτό που ανέφερα προηγουμένως, τα εμπόδια για την πρόσβαση οικονομικά και άλλα εμπόδια για την πρόσβαση στο πολιτισμό. Κύριε Στογεύσκη. Σας ευχαριστώ πολύ, ε, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια παρουσίαση, να σας μιλήσω εδώ για ένα πρόβλημα το οποίο είναι θεμελιώδους ε, σημασίας για την Επιτροπή μας. Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

υπέβαλε, μάλλον παρουσίασε ένα ιδιαίτερο ε, ευρωβαρόμετρο το 399 όσον αφορά την πρόσβαση ε, στον πολιτισμό. Αλλά πέρασαν ήδη πέντε χρόνια σχεδόν. Ε, εκεί είχαμε κάποιες φυγομετρήσεις, είχαμε κάποιες συνεντεύξεις με τους ανθρώπους για να δούμε κατά πόσον συμμετέχουν ή όχι σε πολιτιστικές δραστηριότητες δραστηριότητες και τον τρόπο με τον οποίο ε, κατανοούν τη συμμετοχή στον πολιτισμό. Αυτό ήταν, ε, αυτό ήταν ο κύριος στόχος και και αναδούμε. Ε, αυτοί οι οποίοι ε, δεν συμμετέχουν στις πολιτιστικές αυτές διαδικασίες. Οι περισσότεροι απήντησαν πολύ απλά «δεν με ενδιαφέρει». Όμως δεν έγινε μια προσπάθεια εμβάθυνσης να δούμε δηλαδή για ποιο λόγο υφίσταται αυτό το εμπόδιο, για ποιο λόγο υπάρχει μια δυσκολία πρόσβασης στον πολιτισμό. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να αναφερθώ εγώ στα διαρθρωτικά εμπόδια ε, και στα χρηματοδοτικά εμπόδια ε, όσον αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό. Πρώτο στοιχείο είναι η αναπηρία. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αναπηρία δεν επιτρέπει στους ανθρώπους που από αυτήν υποφέρουν να πάνε στα μουσεία, να συμμετέχουν σε διάφορες εκδηλώσεις κτλ. Δεύτερον, δημοσιονομική διαφορετικές ε, ε, δυσκολίες. Η κάθε χώρα μπορεί να έχει τελείως διαφορετικά φορολογικά συστήματα όσον αφορά τον πολιτισμό και σε ορισμένες περιπτώσεις ε, η φορολόγηση των δραστηριοτήτων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών μπορεί να είναι πάρα πολύ βαριά και μπορεί να είναι και βαριά και η φορολογία για τους ίδιους τους καλλιτέχνες. Τρίτον, ο πλούτος, η οικονομική κατάσταση δηλαδή. Ξέρουμε ότι ε, σε πολλά μουσεία ε, πήραν την απόφαση στη Βρετανία ας πούμε ε, να, είναι, να έχουν ελεύθερη είσοδο αλλά υπάρχουν άλλα μουσεία ε, σε, ε, σε ε, τουριστικές πόλεις, τουριστικά κέντρα λοιπά που έχουν όχι μόνο εισιτήριο αλλά και τσουχτερό εισιτήριο και μάλιστα έχει αυξηθεί πολλές φορές τόσο πολύ η είσοδος που δεν αντέχουν οικονομικά οι επισκέπτες. Υπάρχουν επίσης και ε, εμπόδια ε, τα οποία αφορούν ε, την αδυναμία απορρόφησης του πολιτιστικού προϊόντος λόγω χαμηλού πολιτιστικού επίπεδου και λόγω χαμηλού εκπαιδευτικού επίπεδου για να μπορέσει κανείς ε, να αντιληφθεί ε, την τέχνη και να τον ικανοποιήσει η τέχνη ε, θα πρέπει να έχει ένα βασικό επίπεδο εκπαίδευσης, θα πρέπει να έχει ευαισθητοποιηθεί όσον αφορά την τέχνη και αυτή η ευαισθητοποίηση πρέπει να ξεκινάει από το δημοτικό ακόμα. Επίσης, γεωγραφικά πώς κατανέμονται ε, αυτές ε, οι διαδικασίες, σε ποιες χώρες ε, η κατάσταση είναι καλύτερη, σε ποιες είναι χειρότερη. Εγώ θέλω να καταλάβω γιατί σε ορισμένες χώρες συμμετέχουν περισσότερο τα, οι άνθρωποι σε μουσικές εκδηλώσεις, όπως ας πούμε στη Γερμανία. Ξέρουμε ότι η Γερμανία έχει μεγάλη, μακρά παράδοση όσον αφορά το θέμα αυτό. Ξέρουμε ότι οι Σουηδοί και οι Δανείοι διαβάζουν πολύ, αλλά ε, αυτό δεν συνδέεται ε, με την χρηματοδότηση. Αντιθέτως μάλιστα, ε, ο ΦΠΑ των βιβλίων φαίνεται να είναι πιο υψηλό όσον αφορά τις χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο αναγνωστικό κοινό και χαμηλότερο ΦΠΑ στα βιβλία σε χώρες οι οποίες διαβάζουν λιγότερο. Επίσης πρέπει να ληφθούν υπόψη στο σύνολό του τα στοιχεία αυτά. Η ελλειπή σε συμμετοχή, σε πολιτιστικά, ε, πολιτιστικέ εκδηλώσει κτλ. Υπάρχει ένα τελευταίο στοιχείο ε, Όσον αφορά τους μετανάστες, έχουν, έχουν ληφθεί μέτρα ε, και τα λοιπά, αλλά παρόλα αυτά η προσπάθεια που έχει γίνει έτσι ώστε οι μετανάστες να ενσωματωθούν στις χώρες τις οποίες ε, εγκαθίστανται έχει προκαλέσει κατά κάποιο τρόπο μία έλλειψη αναγνώρισης του πολιτιστικού πλούτου ε, που μπορεί να παρουσιάζουν ε, οι άνθρωποι αυτοί. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει ε, να τα μελετήσουμε όλα αυτά ιδιαίτερα προσεκτικά. Θα σας στείλω τις προτάσεις αυτές όσο γίνεται πιο γρήγορα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις προτάσεις που κάνετε ή θα κάνετε γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι απολύτως απαραίτητες. Το σημαντικό δεν είναι βεβαίως να κάνουμε μονάχα μία διάγνωση του προβλήματος προβλήματος είναι σημαντικό να βρούμε και τον τρόπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσουμε, θα ξεπεράσουμε αυτά τα ε, ε, προβλήματα και τα προσκόμματα τα οποία δεν είναι μόνο υποκειμενικά, είναι και αντικειμενικά. Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Βεβαίως εδώ έχουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Δεν ε, υπάρχουν ισκιώδεις συζητητές σήματα στην αίθουσα. Η Σίλβια. Ναι, ε, αντικαθιστώ εγώ τη συνάδελφο Ροντρίγκε και θα σα διαβάσω αυτά που είχε ετοιμάσει. Οπότε θα διαβάσω το κείμενο. Ε, στον κόσμο όμω ο καθένας βλέπει τον πολιτισμό διαφορετικά. Σήμερα ο κόσμος σέβεται περισσότερο τον πολιτισμό καθώς αντιλαμβάνεται τις δυνατότητες που προσφέρει και που μπορεί να ανοίξει ειδικότερα όσον αφορά τα αποτελέσματα στα κοινωνικά θέματα ενώνει τους ανθρώπους, μειώνει τις ανισότητες. Οι φραγμοί στον πολιτισμό αποτελούν σοβαρό πρόβλημα. Για να τους αντιμετωπίσουμε θα πρέπει να τους συζητήσουμε ευρύτερα από ότι αναφερόμενοι στα απλά καθημερινά εμπόδια ε, συμμετοχή στις πολιτιστικές ε, εκδηλώσεις. Θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα εξισορροπήσουμε την ποιότητα του πολιτισμού και τη βιωσιμότητά του. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, αυτό που με ανησυχεί κυρίως είναι ότι συνήθω δίνεται προτεραιότητα σε άλλους τομείς ε, ει βάρο του πολιτισμού. Ε, τα ευρωπαϊκά προγράμματα όπω το Creative Europe αναγνωρίζει τι δημιουργικέ βιομηχανίε και ότι είναι αναγκαίο να παρασκεθούν επαρκή μέσα για την ανάπτυξή του, διότι αποτελούν κινητήριο δύναμη κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη σε πολλού τομεί. Στο σχέδιο αυτό έκθεση θέλω να συμπεριλάβουμε στρατηγικέ μείωση των δομικών και οικονομικών εμποδίων, Ενδεχομένω μέσω συνεργασίας, παιδείας, ψηφιοποίησης και μέσων. Η παιδεία όχι μόνο μειώνει τα γλωσσικά, φυσικά και γεωγραφικά εμπόδια. Τα μέσα επίσης διαδίδουν τα πολιτιστικά έργα. Τον Ιούλιο του 2017 συζητήσαμε την πρόσβαση στον πολιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκεί οι πολίτε ανέφεραν ότι η έλλειψη πληροφοριών ήταν ο βασικότερο λόγος για τον οποίο δεν συμμετείχαν σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ο κόσμος πρέπει να ενημερώνεται σε σχέση με τα ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί να αξιοποιήσει προ ενίσχυση των ευρωπαϊκών όργων. Επίση, είναι σημαντικό να γίνεται αναφορά στι ε, ε, πιο απομακρυσμένε, ορεινέ περιοχέ. Η πρόσβαση για τους πολίτες αυτών των περιοχών στον πολιτισμό είναι πιο δύσκολη. Η απόσταση, η έλλειψη υποδομών όχι μόνο εμποδίζουν την πρόσβαση σε πολλούς πολιτιστικούς τομείς, διατηρούν επίσης ε, τους πολίτες εν αγνία όσον αφορά τις ευκαιρίες που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ο πολιτισμός έπρεπε να είναι μοχλός όχι μόνο πολιτιστικό, αλλά και για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει για την υποστήριξη των μικρών περιφερειακών οικονομιών ώστε να αναπτυχθεί και μια ευρωπαϊκή ταυτότητα και στι απομακρυσμένες περιοχέ. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε να επικεντρωθούμε και στον εντοπισμό των πιο αδύναμων τομέων του πολιτισμού, να του προβάλλουμε περισσότερο μέσω του ψηφιακού μας θεματολογίου ώστε να γίνουν διαθέσιμοι σε όλους. Το μέλλον της Ευρώπης θα ε, εξαρτηθεί και από την κοινοτομία στον τομέα του πολιτισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Από την Επιτροπή, θέλετε να πάρετε το λόγο. Thank Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Uh, και σας ευχαριστώ και για την πρώτη αυτή ανταλλαγή απόψεων. Κοιτάξτε εδώ, μας ενδιαφέρει η συμμετοχή ε, στην, ε, ε, στον πολιτισμό. Επειδή αναφερθήκατε στο ευρωβαρόμετρο, πρέπει να σας πω ότι μαζεύουμε, συλλέγει η Eurostat στοιχεία και από την έρευνα SILK που αφορά την κοινωνική κατάσταση και ε, ε, ε, τα κοινωνικά στοιχεία έτσι ώστε να δημιουργηθεί έτσι μία ε, πιο ε, συνολική εικόνα. Ε, ίσως μας εκπλήσει το γεγονός ότι σε χώρες με κοινωνικά προβλήματα ή οικονομικά προβλήματα, όπως ας πούμε ήταν η Ελλάδα ή η Ισπανία, δεν προκάλεσε αυτό πρόβλημα όσον αφορά την πρόσβαση στον πολιτισμό. Δηλαδή οι άνθρωποι πηγαίνουν στο σινεμά, πηγαίνουν στο, στα μουσεία. Αυτό που μας προβληματίζει είναι ότι 25% περίπου των Ευρωπαίων Ευρωπαίων απήντησαν λέγοντας ότι δεν συμμετέχουν στις πολιτιστικές διαδικασίες διότι δεν τους ενδιαφέρει. Ε, ε, ε βεβαίως εκεί και η συνειδητοποίηση, η ευαισθητοποίηση αλλά και ε, το εκπαιδευτικό επίπεδο παίζουν σημαντικό ρόλο. Βεβαίως ξέρετε ότι και μέσα από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη προσπαθούμε ακριβώς να ενισχύσουμε αυτούς τους στόχους. Ένας από τους στόχους της προσπάθειας είναι ε, το λεγόμενο non-audience, δηλαδή το κοινό το οποίο δεν ε, μπορεί να το φτάσει ε, και να το αγγίξει καμία πολιτιστική προσπάθεια. Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι του κοινού. Εμείς ε, ε, συμφωνούμε βεβαίως ότι περισσότερες ε, επενδύσεις θα πρέπει να αφορούν την διευρυμένη πρόσβαση εις τον πολιτισμό. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μόργανο. Ευχαριστώ πολύ. Βεβαίω, θα πρέπει να περιμένω να δω τα κείμενα, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι το θέμα αυτό, το οποίο μας απασχολεί σε αυτό το σημείο της ημερησία διατάξεως, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και μας επιτρέπει ω Επιτροπή Πολιτισμού να δούμε λίγο πώς έχουν τα πράγματα όσον αφορά την πολιτική η οποία έχει εφαρμοστεί από το 2014 μέχρι σήμερα ε, σε σχέση με μια πρώτη ας πούμε έκθεση αρκετά ε, πλήρη ε, του συναδέλφου ε, ε, Διακόνου όσον αφορά τον πολιτιστικό πλούτο της Ευρώπης καθώς επίσης και μέχρι την μέχρι το 2018 όπου το Μιλάνο θα είναι πρωτεύουσα της πολιτιστικής οικονομίας της Ευρώπης. Νομίζω ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να περιλάβουμε οπωσδήποτε το θέμα της συμπερίληψης ε, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά τον ρόλο του πολιτισμού. Αυτό είναι ένα στοιχείο λοιπόν το οποίο οπωσδήποτε θα πρέπει με τεπιτάσεως όχι απλά να υποστηρίξουμε αλλά και να προωθήσουμε και να τροφοδοτήσουμε. Κατά αυτή την έννοια λοιπόν έστω και αν δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας νομίζω ότι καλό θα ήταν ε, να επαναλάβουμε τις αρχές που ανέφερε ο συνάδελφος Ζοντεύσκη προηγουμένως ε, ε, και να, να, να λάβουμε υπόψη μας ε, αυτό το στοιχείο του 25% των ανθρώπων που δεν ενδιαφέρονται για, για τον πολιτισμό έτσι ώστε μέχρι το 2018 να μπορέσουμε να έχουμε κάτι επιτυχημένο από άποψη πολιτική και από άποψη πολιτιστική. Ο κύριος για να ολοκληρώσει. Ευχαριστώ, θα είμαι σύντομος. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πάντες εδώ όσους έκαναν παρατηρήσεις. Η Σίλβια Κώστα μίλησε για ένα πολύ σημαντικό θέμα που εγώ δεν είχα αναφέρει. Την έλλειψη ενημέρωσης. Πράγματι, ορισμένες φορές έχουμε ανθρώπους ε, που δεν γνωρίζουν ε, την πολιτιστική προσφορά. Δεν γνωρίζουν τι πολιτιστικές εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα. Επίσης και εγώ θα λάβω υπόψη μου αυτά που προτείνει και η Πρόεδρος ε, ηλική υποδομή. Πρέπει να λαμβάνετε και ηλική υποδομή υπόψη. Καθώς ε, και τις τελευταίες επενδύσεις θα πρέπει να τις δούμε για να καταλάβουμε πού έχουμε ε, πλούσια πολιτιστική προσφορά και για να εντοπίσουμε και τις ελλείψεις. Ευχαριστώ. Πάλι σας ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα μένει να προετοιμάσετε την έκθεση και θα επανέλθουμε τον Ιανουάριο στο θέμα αυτό. Θα ήθελα να σας προτείνω ότι δεν έχει νόημα να είμαστε τρία άτομα εδώ και να πάρουμε το λόγο για το θέμα του Brexit. Ας το αναβάλουμε λοιπόν για την επόμενη συνεδρίαση. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα τόσοι λίγοι να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Αν συμφωνείτε λοιπόν, να περάσουμε στο τελευταίο σημείο της ημερήθειας διάταξης, το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, ακόμα και να είναι τρία μέλη μόνο στην αίθουσα. Σας παρακαλώ πολύ, όποιος δεν ανήκει στο Κοινοβούλιο, να εγκαταλείψουν την αίθουσα, γιατί θα συνεδριάσουμε και κλεισμένο των θυρών. Οπότε θα έχουμε και τον χρόνο, τον απαραίτητο, μέχρι τη συνεδρίαση των συντονιστών. Everyone not part of the European Parliament. Σας παρακαλώ, ποιος δεν ανήκει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκαταλείψει αυτή την αίθουσα.